Je Σας ευχαριστώ παρακαλώ που ήρθατε. Παρακαλώ καθίστε. Παρακαλώ καθίστε, θα ξεκινήσουμε χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση τη συνεδρίασή μας. Δεν θέλω να καθυστερήσουμε γιατί διάφοροι συνάδελφοι θα πάρουν το λόγο στην Ολομέλεια ε, σε λίγο. Επομένως θέλω να προχωρήσουμε γρήγορα. Σας ζητώ να εγκρίνουμε το σχέδιο ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασή μας. Το εγκρίνουμε λοιπόν αφού δεν υπάρχουν αντιρρήσεις και θα ήθελα να κάνω κάποιες ανακοινώσεις. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας μία νέα συνάδελφο, η οποία είναι εδώ παρούσα, η Νόρα Μέμπαρεκ. Καλώς ήλθατε. Καλή δουλειά στην Επιτροπή μας. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι θα πάμε στη Σλοβακία καταληκτική ημερομηνία έτσι ώστε οι ομάδες να ορίσουν τα μέλη που θα συγκροτήσουν την αποστολή είναι σήμερα στη μία η ώρα το μεσημέρι. Επομένως, οι ομάδες που ε, δεν έχουν στείλει ονόματα παρακαλώ να στείλουν στη Γραμματεία για την αποστολή στη Σλοβακία η οποία θα λάβει χώρα το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτά λοιπόν για τις ανακοινώσεις του Προέδρου. Ξεκινούμε την ψηφοφορία. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να έχετε όλοι τις ηλεκτρονικές σας κάρτες, την κάρτα για την ηλεκτρονική ψηφοφορία και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που θέλει να συγχρονίσει τις οικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προωθήσει και να προάγει την ανάπτυξη και τη σταθερότητα, Παρενθετικά, να σας ζητήσω να σοπάσετε παρακαλώ, κάντε λίγο ησυχία, γιατί είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσουμε. Κλείνω την παρέθεση λοιπόν και συνεχίζω λέγοντας ότι σε αυτό το πλαίσιο η Επιτροπή κάθε φθινόπωρο παρουσιάζει έκθεση για τις οικονομικές προοπτικές τη επόμενη χρονιά. Η Επιτροπή Ρέτζι έχει συντάξει γνωμοδότηση από το 2016 κάθε χρόνο με βάση την έκθεση ΕΚΟΝ της Επιτροπής ΕΚΟΝ, ε, της οποία η έκθεση συνδέεται με τον ε, προϋπολογισμό και την ε, κάθε ετήσια οικονομική χρήση. Πάρα πολλές τροπολογίες έχουν υποβληθεί. Ο συνάδελφος εισηγήτρια, η συνάδελφος κυρία Ντονάτο. Μήπως θα ήθελε να πάρει το λόγο πριν περάσουμε στην ψηφοφορία. Αν θέλετε το λόγο τον έχετε, κυρία Ντονάτο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω Ιταλικά. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τη δουλειά που κάναμε μαζί, κυρίως τους κοιόδης εισηγητές και όλους τους βοηθούς, ε, τη γραμματεία, το προσωπικό που μας βοήθησε και είμαι πεπισμένη ότι η γνωμοδότηση που προέκυψε από αυτή την ομαδική δουλειά θα περιλαμβάνει όλα τα βασικά στοιχεία και απόψεις των διαφόρων ομάδων και θα αποτελέσει ένα χρήσιμο έγγραφο προϊόν της Επιτροπής μας ε, προς την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για την ανάλυση και τη βιώσιμη ανάπτυξη του 2020. Νομίζω θα συνεχίσουμε έτσι επικοδομητικά όπως ξεκινήσαμε, τόσο αρμονικά, και στο μέλλον, όπως και για αυτή τη γνωμοδότηση. Σας ευχαριστώ όλους και καλή δουλειά. Ευχαριστώ. Εάν συμφωνείτε λοιπόν, περνάμε ευθύ αμέσω στη ψηφοφορία. Είστε έτοιμοι? Ξεκινούμε με τη συμβιβαστική υπαριθμών 1. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Όχι, συγγνώμη. Διορθώνει ο Πρόεδρος. Πάμε τώρα στην τροπολογία 27. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 48 αποσύρεται. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η συμβιβαστική τροπολογία εγκρίνεται. Περνούμε τώρα στην τροπολογία υπαριθμών 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμ, τροπολογία 101 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται. Τροπολογία 102. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 103. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μπορούμε να υπαλληθεύσουμε την 103 εάν θέλετε. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 103. Πέρας. Εγκρίνεται. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η δική μου κάρτα δεν δουλεύει, δεν λειτουργεί. Καλώς, την 11, συμβιβαστική 11. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβι... Τροπολογία μάλλον 110. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Να το επαληθεψουμε. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 111. Όχι, 110 διορθώνει ο Πρόεδρος. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 110. Πέρας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Την 111 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 113. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 115. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 116. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 117. Υπέρ. Κατά. Αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται. Αλλά μπορούμε να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά εάν το επιθυμείτε. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 117. Πέρασα. Oh. Απορρίπτεται. 118. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. 119. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 120. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Καλώς. Σας υπενθυμίζω ότι θα τα πούμε για την Επιτροπή Ρέτζη στις 19 του μηνός. Σας ευχαριστώ που ήσασταν παρόντες. Ήταν πολύ σημαντική η μερίσια διάταξή μας και θα ήθελα να κάνω κάποιες ανακοινώσεις για την πρόοδο των νομοθετικών φακέλων που μας αφορούν και πιο συγκεκριμένα το Ταμείο για τη Δίκαιη Μετάβαση. Καλή Ολομέλεια. Θα τα πούμε τότε στις 19 του μηνό για τη συνεδρίασή μας. Ο Πρόεδρος ευχαριστεί τους διερμηνείς και το προσωπικό και εμείς. Ah, quel est son nom Bien, je n'avais pas euh, noté. Δεν είχα παρατηρήσει την παρουσία σας. Έχουμε ένα νέο μέλος. Δύο νέα μέλη. Βιτσέζο Σόφο και την κυρία Τζέμα. Προφανώς και σας καλωσορίζω. Καλώς ήλθατε. Ελπίζω ότι θα συμβάλλετε στις εργασίες της Επιτροπής μας. Ελπίζω να τα ξαναπούμε στις 19 να σας δούμε για τις εργασίες της Επιτροπής μας, οπότε και θα κάνω τις ανακοινώσεις που σας είπα. Καλώς ήρθατε και πάλι. Συζητώ συγγνώμη που δεν σας είδα. Η κυρία Ντονάτα θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και περνάω στα Ιταλικά. Είμαι απογοητευμένη από την αρνητική ψήφο. Δεδομένου ότι οι περισσότερες ε, τροπολογίες ε, εγκρίθηκαν και υπήρχαν και πολλές τροπολογίες που είχαν συμπεριληφθεί. Και είναι κρίμα, γιατί η δουλειά ήταν πολύ επικοδομητική, πολύ αρμονική η δουλειά που έγινε δηλαδή με τους συναδέλφους και τους εισηγητές. Υπάρχει ένα θέμα πολιτικό εδώ, απέναντι στην ομάδα μας πια. Πέρα από το περιεχόμενο, πέρα από τη δουλειά που κάνανε τα επιμέρους οι επιμέρους βουλευτές πάνω σε αυτή την έκθεση. Είναι θλιβερή αυτή η κατάσταση. Θέλω να το υπογραμμίσω. Δεν νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δουλέψει αποτελεσματικά αυτή η Επιτροπή. Το καταγράφω αυτό. Ευχαριστώ όμως όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί μου και έδειξαν την εκτίμησή τους, με στήριξαν. Ελπίζω κάποια στιγμή αυτή, αυτός ο υγειονομικός αποκλεισμός να σπάσει και να πριτανεύσει λογική επιτέλους. Να υπάρξει θετικό πνεύμα, επικοδομητική διάθεση και κυρίως σεβασμός της δημοκρατίας. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας και τώρα κλείνουμε τη συνεδρία.